ευρύτερη πληρέστερη στρατηγική για να προωθήσουμε ένα πιο ισοδίκαιο, υγιέστερο και πιο ειρηνικό πλανήτη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Μάρτιν. Για την Επιτροπή Ανάπτυξη έχουμε δύο μιλητέ. Καταρχήν ο κ. Κατσμαρέκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ.